Ε, για τα σχόλιά σας. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση στο θέμα αυτό και τώρα και ευχαριστώντας τους ε, παρεμβαίνοντες Θέλω να σας ενημερώσω τώρα δυνάμει του άρθρο 131 του κανονισμού μας ότι οι διορθώσεις δεν κατατέθησαν εχθές αυτό σημαίνει ότι εγκρίνονται τα κείμενα όπως διορθώθηκαν. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έκθεση προόδου